Good morning, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε. Τη συνεδρία τη Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα, στι ανακοινώσεις ε, της Προέδρου, κάποια ζητήματα. Καταρχήν, σήμερα 11 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής Μέρα των Κοριτσιών Πολλές φορές έχουμε μιλήσει εδώ για τα μικρά κορίτσια, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την καταπολέμηση της οικιακής βίας και βεβαίως το θέμα της α, ε, μια σειρά αποζητήματα λοιπόν που μας έχουν απασχολήσει. Ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στη σημασία αυτής της μέρας και για τα κορίτσια αυτά και για μας. Να σας πω επίσης ότι στις 13 Οκτωβρίου στις 10, 10 με 11 το πρωί θα λάβατε σχετικό mail θα γίνει μια εκδήλωση με την πρώην πρόεδρο της Σρι Λάνκα την κυρία Βαντάρα Νάικε Βανταρανάη και Κουμπαρατούγκα, ελπίζω να το πρόφερα σωστά. Την έχουμε καλέσει για να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση. Έχετε λάβει τις σχετικές πληροφορίες και ελπίζω να είστε εκεί. Και μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης. Ψηφοφορίες. για το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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές λοιπόν να το επαληθεύσουμε αυτό το δεύτερο μέρος τροπολογίας 3 λοιπόν ψηφίζουμε πέρα. <laughs> Se abre, se abre la votación. Se cierra. Peras psiforías. Κάποιος αντιπρόεδρος δεν είχε την κάρτα μαζί του. Εν πάση εγκρίνεται η τροπολογία 10 υπέρ 9 κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, λάθος. 11 υπέρ, 9 κατά. Έτσι λοιπόν εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. Πολύ ωραία. Και μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. τροπολογία, ε, μάλλον ε, κείμενο για την ε, ισότητα των δύο φύλων στις εμπορικές συμφωνίες.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 Eh, Συνεχίζουμε λοιπόν με την εμείς διάταξη το σημείο 11 ισότητα των δύο φίλων στις εμπορικές συμφωνίες. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Φοντάνα η οποία θα κάνει σχετική παρουσίαση. Πρόκειται για μια μελέτη την ανάλυση από τη σκοπιά των δύο φίλων σε ό,τι αφορά την συμφωνία ΣΕΤΑ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Ευχαριστούμε την κυρία Φοντάνα που συμμετέχει σήμερα στη συζήτηση. Έχετε το λόγο για την παρουσίασή σας και στη συνέχεια βεβαίως να γίνει μια συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα και βεβαίως αναμένω τα ερωτήματά σας, τα σχόλιά σας που σίγουρα θα βελτιώσουν την ποιότητα του τελικού εγγράφου. Μου ζητήθηκε να κάνω μια αξιολόγηση για το κατά πόσο οι εμπορικέ συμφωνίε που είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνουν επαρκή σημασία στου στόχου περισσότερων των δύο φύλων. Μια σειρά από συμφωνίε αυτή τη στιγμή ε, είναι υποδιαπραγμάτευση. Η συμφωνία ΣΕΤΑ, η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά, το TTIP με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η εμπορική συμφωνία στον τομέα των υπηρεσιών που αφορά πολύ περισσότερες χώρες. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σήμερα ιδιαίτερα στο ΣΥΕΤΣΕΤΑ διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι έχω καταλάβει θα πρέπει να πάρει μια απόφαση για το κατά πόσο θα εγκρίνει την ΣΕΤΑ εντό των επόμενων εβδομάδων. Πολλά από τα σημεία, πολλά από τα σχόλια που θα κάνω σήμερα ε, έχουν σημασία και για τις λοιπές συμφωνίες όμως, ισχύουν και τις λοιπές συμφωνίες. Αυτές οι συμφωνίες ε, αποτελούν μέρος ε, μιας νέας γενιάς εμπορικών συμφωνιών με την έννοια ότι δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών, περιλαμβάνουν υπηρεσίες, επενδύσεις, άλλους τομείς που σχετίζονται με το εμπόριο, πνευματική ιδιοκτησία, δημόσιες προμήθειες κτλ. Όλες αυτές οι πτυχές θα έχουν ενδεχομένως σημαντικές επιπτώσεις σε τις σχέση των δύο φύλων ε, και πρέπει να τις ερευνήσουμε διεξοδικά. Η πρώτη γρήγορη απάντηση στο ερώτημα ε, του κατά πόσο τα ζητήματα ισότητας δύο φύλων λαμβάνονται υπόψη είναι όχι. Αυτή είναι η απάντηση, η απλή. Η ισότητα των δύο φύλων σε τέτοια ζητήματα εξετάζεται σε ένα πολύ στενό πλαίσιο ε, η απασχόληση σε συγκεκριμένους ε, κλάδους δεν γίνεται μια ανάλυση σε ευρύτερες πτυχές. Οι επιπτώσεις ε, των εμπορικών συμφωνιών στα ζητήματα ισότητας των δύο φύλων είναι όμως πολύ ευρύτερες. Χρειάζεται λοιπόν μια συστηματική προσέγγιση, διότι το εμπόριο ποτέ δεν είναι ουδέτερο σε ό,τι αφορά τα δύο φύλλα. Διότι οι οικονομικές δομές ε, εντός των οποίων λαμβάνει χώρα το εμπόριο έχουν δημιουργηθεί με βάση την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια βιώσιμη αξιολόγηση αντικτύπου της ΣΕΤΑ που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κάνω κάποιες συστάσεις αξιολόγησης και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ ε, στην ε, σημαντική βιβλιογραφία που υπάρχει ε, για τα θέματα αυτά για να βρούμε κάποια συστατικά στοιχεία να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να μπορεί να μα επιτρέψει να αναλύσουμε τα θέματα ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην εμπορική πολιτική και θα αναφερθώ επίσης ε, στην ανάγκη μιας ισχυρότερη παρουσίας του ζήτηματο αυτού στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση ε, για το ΣΕΤΑ. Θα ε, σα πω τι καλύπτει το ΣΕΤΑ αυτή τη στιγμή, τι δεν καλύπτει, τι θα έπρεπε να καλύπτει και τέλο θα αναφερθώ στο γεγονό ότι πρέπει να δεσμευτούμε ε, να εξετάσουμε ζητήματα ισότητα φύλων σε διάφορε φάσει διαπραγμάτευση, ήδη από τη φάση διαβούλευση, στην αρχή δηλαδή. Ποια είναι τα βασικά συστατικά μια ανάλυση ε, εμπορική και ισότητα των δύο φύλων. Η βιβλιογραφία για το ζήτημα αυτό δεν είναι μεγάλη. Υπάρχει μια διάδραση μεταξύ ε, ισότητας φύλων και εμπορίου το εμπόριο υπό τις διάφορες μορφές του ε, επηρεάζει τα δύο φύλλα ε, και τούμπαλιν. Όταν μιλάμε για gender, βέβαια, τα δύο φύλλα ε, πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε. Είναι πολλοί τρόποι επιρροής, επίδρασης. Ε, και οι άντρες και οι γυναίκες είναι παραγωγοί, είναι εργαζόμενοι, είναι καταναλωτές. Είναι πολίτες, είναι φορολογούμενοι, οι οποίοι ε, δικαιούνται πρόσβαση σε μια σειρά από δημόσιε υπηρεσίε. Το εμπόριο λοιπόν επηρεάζει την απασχόληση. Αυτό συνήθω ε, ε, ακούμε. Αλλά είναι σημαντικό για να καταλάβουμε όχι μόνο τι συμβαίνει σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων εργασία, αλλά και με την ποιότητα των θέσεων αυτών. Το εμπόριο επίση επηρεάζει και την κατανάλωση διότι αλλάζει τις τιμές των αγαθών, των διαθέσιμων αγαθών και μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις για τα δύο φύλλα, ε, για την ισότητα των δύο φύλων. Παραδείγματος χάρη συχνά η ευθύνη για την αγορά των τροφίμων αλλά και, την, ε, και το μαγείρεμα ε, είναι συχνά των γυναικών. Στα πλαίσια των νέων εμπορικών συμφωνιών που περιλαμβάνεται η απελευθέρωση των υπηρεσιών, οι προμήθειες κτλ. Ε, υπάρχει το θέμα των του δημόσιου σκέλους. Απελευθέρωση των υπηρεσιών ε, μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα που έχει μια κυβέρνηση να παράσχει υπηρεσίες. Μπορεί να αλλάξει η σύσταση ε, των κυβερνητικών δαπανών και αυτό θα έχει επιρροές, θα, θα επιδράσει τα δύο φύλλα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για υπηρεσίες που συνήθω ε, δημόσιες πολιτικές, υπηρεσίες και πολιτικές που υποστηρίζουν τι γυναίκε ε, στον τομέα της περίθαλψης, ε, της υγείας. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά. Δεν υπάρχουν, όπως είπα, πολλά βιβλιογραφικά στοιχεία από αυτού, αλλά το γεγονό ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιπτώσει για τα δύο φύλλα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν οι έρευνες εδώ. Το αποτέλεσμα λοιπόν της απελευθέρωσης του εμπορίου είναι περίπλοκο, είναι αντιφατικό και δεν αφορά μόνο άντρες και γυναίκες. Θα υπάρξουν διαφορές μεταξύ διαφόρων ομάδων γυναικών, μεταξύ ε, γυναίκες που δουλεύουν στα εργοστάσια και γυναίκες που δουλεύουν ε, ε, στον αγροτικό τομέα. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην κατανομή της εργασίας, ε, της, πλη, της πληρωτέας εργασίας, αλλά και της εργασίας η οποία δεν πληρώνεται. Έγινε λοιπόν μια αξιολόγηση για τη ΣΕΤΑ ε, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βιώσιμη μελέτη δικτύπου χρησιμοποιείται από το 1999 ως ένα μέσο για να αξιολογούμε τις ε, κοινωνικές, περιβαλλοντικές ε, επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών. Η πρόθεση είναι αυτό να είναι ένα βασικό εργαλείο για να καλυφθούν και τα ζητήματα ισότητας των δύο φύλων. Ένα πολύ καλό έγγραφο το οποίο προετοιμάζει η Βίλουπ δείχνει ότι η κάλυψη των ζητημάτων ισότητας των δύο φύλων ε, ποικίλει. Και ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχω κάνει μια ανάλυση κειμένου της έκθεσης, 500 σελίδες βέβαια είναι αυτή η έκθεση και οι γυναίκες και στους δύο φίλους αναφέρονται μόλις δύο φορές στις 500 σελίδες. Από ό,τι φαίνεται, μάλιστα αυτό που, συμβαίνει, ε, η επιπτώσει για τους άντρες δεν υπολογίζονται όσο ότι επηρεάζουν τις των δύο φίλων. Παραδείγματος χάρη στον τομέα ε, των ορυχείων, ε, εφόσον λέει η έκθεση κυρίως εργάζονται άντρες στον τομέα αυτών, τον εξορυκτικό, ε, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις για την ισότητα των δύο φύλων. Και... Λες και η ισότητα των δύο φύλων εξαρτάται μόνο από το τι θα γίνει με τις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές ε, προβολές που γίνονται, ε, είναι ένα μοντέλο πολύ συγκεκριμένο περισσορροπίας των δύο φύλων στις προσωμιώσεις αυτές και υπάρχουν πολύ λίγες μεταβλητές. Από ό,τι φαίνεται όλα έρχονται να προσταθούν στη συνέχεια. Δεν, δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται από την αρχή της την ανάλυση δηλαδή. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το, περιορισ... το, το, πόσο περιορισμένη αυτή είναι η προσέγγιση του συγκεκριμένου μοντέλου. Διότι έχω συνεργαστεί με το μοντέλο, το μοντέλο του CGE τα τελευταία χρόνια. Ε, πριν από 15 χρόνια ε, προετοίμασα το πρώτο CGE μοντέλο που να, που να λαμβάνει υπόψη την ισότητα των δύο φύλων. έχουμε αποδείξει ότι μπορούν στοιχεία που φέρνουν στο δύο φύλων να συμπεριληφθούν στο μοντέλο από την αρχή. Έχει ξαναγίνει κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο Μπαγκλαντές, στη Ζάμπια και βεβαίως είναι κάτι που μπορεί να γίνει και σε χώρες όπως ο Καναδάς και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα στατιστικά στοιχεία για τον δύο είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια δικαιολογία να πούμε ότι είναι περίπλοκο. Όχι, αυτά τα μοντέλα μπορούν να ενσωματώσουν την προσέγγιση ισότητας των δύο φύλων. Υπάρχει μια τομεακή ανάλυση λεπτομερής, αλλά δεν αναφέρεται η επιπτώσεις ό,τι αφορά την κατανομή εντός της κάθε χώρας. Και είναι σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε ποια δυναμική μπορεί να ενεργοποιηθεί ε, από μια τέτοια εμπορική συμφωνία. Δεν έχουμε λάβει δηλαδή στοιχεία στο μοντέλο αυτό σχετικά με τους κερδισμένους και τους χαμένους εντός της κάθε χώρας της Ένωσης. Αναφύλλω, ε, ανα τύπου νοικοκυριού, ανα ε, τομέα εργασίας. Είναι σημαντικό όμως να το δούμε αυτό και να δούμε ποια συμπληρωματικά μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να προστατεύσουμε ευάλωτες ε, ε, κατηγορίες ανδρών και γυναικών που θα επηρεαστούν. Και αυτό ευθυγραμμίζεται με τη νέα αρχή του να προωθήσουμε πολιτικές που δεν αφήνουν κανένα πίσω, όπως ε, λέει η ατζέντα για την βιώσιμη ανάπτυξη του 2030. Βεβαίω, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στον οικονομικό αντίκτυπο, αλλά πρέπει να δούμε και άλλου τύπου αντικτύπου, ποιοτικέ ε, επιπτώσεις, να μην αναφερόμαστε μόνο σε ποσοτικά στοιχεία. Ποιε είναι οι βασικέ συστάσει τώρα, τι οποίε έχω αναπτύξει βεβαίω πολύ ευρύτερα στον έγγραφο, για να ενισχυθεί η, ε, η σημασία της όρτας των δύο φύλων στην αξιολόγηση. Καταρχήν πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, στοιχεία που αφορούν τα δύο φύλλα, στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε στοιχεία ε, τα οποία να μας βοηθούν να καταλάβουμε ποια θα είναι η δυναμική σε ό,τι των δύο φύλων. Έχουμε στοιχεία, παραδείγματο χάρη, για την πρόσβαση των οικοκυριών στις υπηρεσίε, στις κοινωνικέ υποδομέ, που μπορούν να μα βοηθήσουν να καταλάβουμε τη δυναμική που δημιουργείται ακόμα και αν δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ε, αναφύλω. Να προσπαθούμε πάντως να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους στατιστικά στοιχεία αναφύλω σε όλη την ανάλυση. Επίσης να εξετάζονται όχι μόνο αριθμοί, αλλά και τις, ε, τους κανόνες. Να καταλάβουμε δηλαδή αν υπάρχουν αλλαγές στην ποιότητα ε, της εργασίας, στις συνθήκες εργασίας ε, και λόγω των χαρακτηριστικών αυτών των νέων εμπορικών συμφωνιών είναι κρίσιμη σημασία να καταλάβουμε καλύτερα τι επιπτώσει για τα δύο φύλλα της, ε, του εμπορίου των υπηρεσιών και τι ενδεχόμενε αλλαγέ ό,τι αφορά την ποιότητα και την πρόσβαση ε, στην, στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτά είναι τα σημεία κλειδιά για την ενίσχυση της ανάλυσης. Υπάρχει όμως και μία ανάγκη να ενισχύσουμε και τη δέσμευση απέναντι στην ανησυχία ε, στην προβληματική των δύο φύλων, στις διαπραγματεύσεις αυτές. Πρέπει οι, οι ομάδες γυναικών να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αλλά δεν αρκεί. Εάν δεν υπάρχει κανεί στην βασική ομάδα έρευνα που να είναι ειδικό στα ζητήματα των δύο φύλων, είναι αρκετά απίθανο οι ανησυχίε που τίθενται από ομάδε γυναικών να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση. Η σύστασή μου λοιπόν είναι, διότι υπάρχουν εμπειρογνώμονε, να υπάρχουν εμπειρογνώμονε για ζητήματα των δύο φύλων στην ομάδα, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι εμπειρογνώμονε για τα πάντα βέβαια, οπότε καλό θα είναι να είναι δύο. Ένα οικονομολόγο και κάποιος που να έχει ε, κάνει έρευνα σε άλλους ε, τομείς κοινωνικών επιστημών. Εξέτασα τον κατάλογο των ερευνητών που συμμετέχουν στην ομάδα παξιολογή της τη ΣΕΤΑ. Γνωρίζω μάλιστα κάποιους από αυτούς. Είναι νέα τα μέλη και είναι όλοι άντρες. Και βεβαίω δεν υπάρχει εμπειρογνώμονα ειδικό σε αισθήματα σώτα των δύο φύλων. Είναι σημαντικό λοιπόν όχι μόνο να υπάρχει πραγματογνωμοσύνη στην ομάδα έρευνα για τα στήματα ισότητα των δύο φύλων, πρέπει επίση να υπάρχει μια τακτική κατάρτιση των αξιωματούχων, των διαπραγματευτών. Ε, υπάρχουν πολλά καλά εργαλεία, πλαίσια, υλικό εκπαίδευση και κατάρτιση που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και έχω συνεισφέρει ε, σε πολλά από τα προγράμματα κατάρτισης αυτά το τελευταίο από αυτά έγινε από την UNTAC, είναι δύο, από την UNCTA μάλλον, είναι δύο τόμοι, ε, εξαιρετικοί. Υπάρχουν και άλλες ε, πηγές. Υπάρχει υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως περιπτώσει, έτσι ώστε να προωθηθεί η συμπερίληψη, η μεγαλύτερη συμπερίληψη των ζητημάτων σε όλους των δύο φίλους διαπραγματεύσεις. Αυτά είχα να σας πω και αναμένω τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φοντάνα και τώρα αρχίσουμε τον γύρο των ερώτα απαντήσεων. Η κυρία Νόελ πρώτη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τους παρουσιάσεις. Ήταν άντρες και αυτοί που εξελόγησαν αυτά τα έγγραφα ή τα προετοίμασαν και εμένα θα με ενδιαφέρει προσωπικά. Γιατί αφορά μια ενδιάμεση μελέτη για το αν περιλαμβάνονται σε εμπορικέ συμφωνίε ε, η πτυχή του φύλου. Κατά την άποψή μου, στατιστικά δεν έχει αποδειχθεί ποιε επιπτώσει θα έχει η ΣΕΤΑ. Θα έχει συγκεκριμένα στι γυναίκε τη Ευρώπη και στι γυναίκε και στου άντρε ε, του Καναδά δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη δήλωση για το πώς θα, ε, επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων και των γυναικών και παράλληλα δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα που να βοηθήσει τη σύναψη της συμφωνίας. Δεν υπάρχει η οπτική προς το μέλλον. Και τρίτον, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, το είπατε στην πρώτη σας ε, πρόταση, ότι είναι μια νέα συμφωνία μια συμφωνία που δεν έχει να κάνει μόνο με προϊόντα αλλά και με υπηρεσίες. Και επομένω αυτή η νέα γενιά συμφωνιών πιστεύετε ότι, ότι τέτοιου είδου συμφωνίες θα έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες από ό,τι άλλες συμφωνίες. Ειδικά όσον αφορά το δημόσιο τομέα ο οποίος είναι, ε, στον οποίο εστιάζει αυτή η νέα συμφωνία. Ευχαριστούμε κυρία Νόηλ. Κύριε Ρούτασον έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την ε, εισήγησή σας και είναι πάρα πολύ ανησυχητικά όλα αυτά τα οποία μας εξηγήσατε για το τι γίνεται με αυτές τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Πάντως, να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ένα από τα θέματα μας έχουν απασχολήσει όταν αξιολογήσαμε αυτές τις συμφωνίες ήταν το μοντέλο CGA όσον αφορά τις επιπτώσεις για την απασχόληση και είπαμε ότι δεν είναι αξιόπιστα τα δεδομένα ε, ευτυχώς για το, τη συμφωνία ΣΥΤΑ ε, ε, χρησιμοποίησαμε άλλα μοντέλα και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε και εσείς για το μοντέλο αυτό το CGA αν μπορείτε, πέστε μας δύο λόγια παραπάνω. Έχει χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού η αξιολόγηση κάποια συμφωνίας. Κυρία Αρένα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και συμμερίζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων και όχι μόνο όσον αφορά την προσέγγιση ανά φίλο ή την προσέγγιση χωρίς ανάλυση δεδομένου αναφύλου. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται αν υπάρχει κέρδος ή ζημία από αυτές τις ε, συμφωνίες με βάση το μοντέλο ΣΕΖΕ και τελικά είναι δύσκολο να γίνει η ανάλυση των αρνητικών. Όλοι λένε ότι σε τέτοιου περιπτώσεις μέτρων επί τη βάση της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν τα θετικά, αλλά υπάρχουν και τα αρνητικά για κάποιους άλλους. Οπότε θα πρέπει να παρασκευαστούν κατά κάποιο τρόπο οι Ευρωπαίοι για αυτό το σοκ της παγκοσμιοποίησης ε, να βρούμε επομένω κάποιο μοντέλο το οποίο ανά χώρα και ανακλάδο της οικονομίας να μας παρουσιάζει τα αρνητικά και έτσι να μπορούμε να δουλέψουμε σωστότερα όταν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Τι γίνεται, βλέπουμε αυτές τις ε, συμφωνίες ε, εμπορίο, με Καναδά, με ΙΠΑ, με το Μεξικό και δεν έχουμε κάποιες ε, μελέτες, έστω και αυτές όπως το ΣΕΖΕ που αμφισβητούνται. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποιες άλλες ε, συμφωνίες από πλευράς φίλων. έχουν κάποιες συμφωνίες 20 ετίας, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευράς αυτών των συμφωνιών, το TTIP, τη ΣΕΤΑ, για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον κόσμο. Αλλά από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν μας τα δίνουν. Να δούμε ακριβώς τι έγινε αυτή την 20 ε, ετία. Εκεί, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού επίσης, μας είπατε για ΣΕΤΑ, TTIP, ΤΙΖΑ, ε, ε, τις συμφωνίες Βορρά με το Βορρά. Δεν μας είπατε τι γίνεται με αυτές τις συμφωνίες τερικής σχέσης Βορρανότου, όπως ας πούμε με την Αφρική. Ε, θα συζητούμε τώρα εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί και εκεί υπάρχουν επιπτώσεις όσον αφορά τα δύο φύλλα. Όχι μας μόνο στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα σε όλο τον κόσμο. Για πες μας τι γίνεται με αυτές τις ε, συμφωνίες ομένως οικονομικής συνεργασίας. Κυρία Μπιόρκ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Θέλω κάτι να πω στις στην συνέχεια των όσων είπε η συνάδελφο. Τι γίνεται με κάποιες εμπορικέ συμφωνίες. Μπορούμε να κάνουμε κάποια ανάλυση όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσει, τι κρατικέ, υπηρεσίες. Πώς επιδρούν αυτές ε, στις, στη ζωή των γυναικών, στην ισότητα των φίλων. Τι γίνεται με αυτές τις συμφωνίες. Βέβαια, στις 18 Δεκάτου θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Άρα Τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, αλλά τι γίνεται τέλο πάντων με τις πιο πρόσφατες συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Τι γίνεται εκεί με την ισότητα των φίλων, κυρία Κολόμσκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλους και όλες που έλαβαν τον λόγο. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών για τις γυναίκες, να λάβουμε υπόψη τα γενικά χαρακτηριστικά αυτών των συμφωνιών. Και έτσι θα δούμε πώς ε, επηρεάζονται οι γυναίκες. Τι γίνεται με την αγορά. Η ΣΥΤΕΠΑΜ θα φέρει απορρίθμιση στην αγορά, θα γίνει πιο ανοιχτή η αγορά. Όμως αυτή η αγορά θα είναι καλύτερη για τις γυναίκες ή όχι. Να, ποιες διαφορές θα πρέπει να αναζητήσουμε. Μήπως και τα πράγματα γίνουν χειρότερα για τις γυναίκες. Μήπως οι γυναίκες ε, χρειάζονται κάποια εργαλεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, για να μπορέσουν να κινηθούν στη βάση της ισότητας με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην αγορά. Γκέρικ. Όσον αφορά τι νέε συμφωνίε, ε, πρέπει να πω ότι τι παλιές ούτε καν ελέγξαμε. Υπάρχει ένα ειδικό ρόλο εδώ. Υπάρχουν ε, στην Ισπανία όμιλοι επιχειρήσεων που αναλύουν τον ρόλο των γονέων και που ε, ορίζουν και κανόνες. Υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε γονείς και σε οικογένειες χωρίς παιδιά ε, σε αυτή την ανάλυση που κάνατε. Bueno, finalizado este turno de intervenciones. Eh. Ολοκληρώθηκε αυτό ο γύρο ερωτήσεων. Κύριε Φοντάνα, έχετε το λόγο για να τι απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω καταρχά πόση ώρα έχω για να απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα. 15 λεπτά. Θα κάνω επιλογές, λοιπόν. Θα απαντήσω επιλεκτικά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα ερωτήματα, τα βασικά τουλάχιστον γιατί κάποιοι άλλο καλύπτονται κιόλα. Κατά πρώτον, υπάρχουν στατιστικές και πολλές ε, που αναλύουν βάση το φύλλο σε εθνικό επίπεδο ε, στην Ευρώπη καθώς και στον Καναδά. Απλώς αυτές οι στατιστικές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για να αναλύσουν τον αντίκτυπο ε, στο εμπόριο άρα δεν έχουν σωματωθεί στο μοντέλο το οποίο ανέφερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί πίνακες που αφορούν την απασχόληση σε αυτή την ε, έκθεση, αλλά αυτή είναι μια κατηγορία η οποία όταν κάνουν κάνει διάκριση ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Έχουμε πολλές στατιστικές και κάτι για το οποίο ανησυχώ είναι ότι κάνουμε λόγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στην Ευρώπη στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε τις διαφορές ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Η Γεωργία θα επηρεαστεί από την ΣΕΤΑ στη Ρουμανία. Το 35% των γυναικείων εργασιών είναι στην Γεωργία, στη Γερμανία, στην Δανία και σε άλλες χώρες. Από εκείνη την πλευρά μόνο το 1% των αγροτικών εργασιών αφορά τις γυναίκες. Άρα οι γυναίκες στη Ρουμανία θα επηρεαστούν περισσότερο. Αν υπάρχει κάποια επιρροή στην Γεωργία. Επίσης γνωρίζω διάφορες εργασίες που έχουν διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τα μέτρα λιτότητας όπου δεν μελετά τον αντίκτυπο στο εμπόριο αλλά τον αντίκτυπο σε σχέση με το φύλλο στις ε, κοινωνικές δαπάνες και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον όπου θα μπορούσαμε να αναλογιστούμε ποιες θα ήταν οι ε, Και αυτό απαντάει και το ερώτημα για το αν λαμβάνουμε υπόψη τους γονείς, τα άτομα παιδιά. Οι περικοπές αυτές ε, πρέπει να δούμε ποιους επηρεάζουν πιο αρνητικά. Μονογονικές οικογένειες, ε, μητέρες με παιδιά και χαμηλοσυνταξιούχους. συνταξιούχους. Πολλές από αυτούς είναι γυναίκες, είναι χείρες, γιατί συνήθως ζουν περισσότερο από τους άντρες και χρειάζεται να αγωνιστούν γιατί έχουν ακριβώς χαμηλότερες συντάξεις. Όταν υπάρχει υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών, τότε οι πιο ευάλωτες κατηγορίες γυναικών θα επηρεαστούν Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει ανάλυση όχι μόνο ανάλογα με το φύλλο αλλά και ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, το μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τα δεδομένα υπάρχουν, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Μπορούμε να κάνουμε πολλά με τα υπάρχοντα δεδομένα. Τη ονομάζω μια νέα γενιά συμφωνιών. Δεν είναι ακριβώς μια νέα γενιά συμφωνιών, γιατί η πρώτη συμφωνία που ε, υπερεύαινε ε, τα αγαθά και είχε να κάνει και με επενδύσεις και εμπόρια ήταν η ναύτα το 1999. Όμως αυτή η έννοια της απελευθέρωσης ε, των υπηρεσιών, των δημόσιων δαπάνων είναι πιο έντονη σε αυτές τις συμφωνίες. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις στην κατανομή και στο φύλλο, όμως δεν υπάρχει αρκετή τεκμηρίωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση και να προωθήσουμε την έρευνα για να καταλήξουμε συμπεράσματα. Υπάρχουν έργα που έχουν γίνει τελευταία χρόνια από ερευνητέ και ομάδες γυναικών για την επίπτωση της ε, λιτότητας στην Ευρώπη, τα οποία μπορούν να μας ε, βοηθήσουμε να καταλάβουμε. Ακόμα και το μοντέλο CGE. Να σας εξηγήσω προς αυτό. Ε, με είχαν καλέσει σε, ένα, σε μια συντηρηστησία το 2000 για να παρουσιάσω το έργο μου, όμως δεν ε, δόθηκε συνέχεια σε αυτό. Έχω εργαστεί για τη Ζάμπη, για το Πακιστάν και έχω κάνει αναλύσεις και έχω εκδώσει αυτό το βιβλίο που ονομάζεται «Η φεμινιστική πτυχή στο εμπόριο». μου ζήτησαν να δω ποια θα είναι η επιπτώση της, ε, στις στο TTIP. Όμως η εμπειρία μου είναι κυρίως στις ε, εμπορικές πολιτικές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2009 κάναμε μια αξιολόγηση της επίπτωσης σε τρεις, σε τρεις χώρες, στην Τανζανία. Επιλέγαμε μία ε, χώρα από κάθε γεωγραφική ομάδα. Και μελετήσαμε την επίπτωση της απελευθέρωσης των αγαθών και αφορούσε και το γεγονός ότι εξαρτώνταν πολύ από του ε, τους προ τα ε, εθνικά έσοδα. Στη Μοζαμβίκη λοιπόν α, ε, διαπιστώθηκε ότι θα υπάρξει μείωση στα έσοδα από τους δασμούς και ότι αυτό θα οδηγούσε σε περικοπές, σε κοινωνικά προγράμματα Κάτι που θα ήταν πολύ καταστροφικό για τις γυναίκες. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες, υπάρχουν μελέτες για το αντίκτυπο στην κατανομή, κατανομή στην ναύτα και αυτό το αναφέρω στο τελικό έγγραφο για τα μαθήματα που μπορούμε να αντιλήσουμε από αυτό Όμω πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι συνθήκε είναι διαφορετικέ σε αυτέ τι τρει νέε συμφωνίε. Γιατί οι συμφωνίε είναι μεταξύ βορρά και βορρά, γιατί η ναύτα ήταν σε άλλο επίπεδο προφανώ, σε διαφορετικό αναπτυξικό επίπεδο μεταξύ των δύο εταίρων. Άρα κάτι διαφορετικό θα συμβεί εδώ. Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία, έχουμε τα δεδομένα, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι ερευνητές, και εμπειρογνώμονες που θα προσπαθήσουν να μελετήσουν σε βάθος όλα αυτά. Συμφωνώ. Συγγνώμη, δεν προθυμηθώ όλα τα ονόματά σας, αλλά είναι σημαντικό όντως να καταλάβουμε ποιες είναι οι επιλογέ όλων των αλλαγών που θα λάβουν χώρα. Ε, τη της και άλλες πτυχές. Είναι σημαντικό όχι μόνο να απορρίψουμε τις συμφωνίες αυτές, αλλά να έχουμε επίγνωση της επιπτώσης στο φύλλο και να σκεφτεί κάθε χώρα συμπληρωματικά μέτρα για να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες. Γιατί αν δούμε ότι οι θα είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν θα οδηγηθούμε στο να απορρίψουμε κατευθείαν τι συμφωνίε αυτέ. Δεν ξέρω αν κάλυψα τα ερωτήματά σα, όμω είμαι διαθέσιμη και για περαιτέρω ερωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φοντάνα, λέει η πρόεδρο. Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μα πάνω στο θέμα αυτό, γιατί πραγματικά μα ενδιαφέρει γι' αυτό και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα δηλαδή τι γίνεται όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και την ισότητα των φύλων. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Και σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημέρα σε διάταξη. Είναι η έκθεση για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 14 έως 15. Ο κύριος Κορτάσον είναι ο εισηγητής. Χτες για το ίδιο ζήτημα είχαμε την ακρόαση. Σήμερα θα ακούσουμε την εισήγηση του συντάκτη της έκθεσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και χτες είχαμε εκείνο το εργαστήριο και την σχετική συζήτηση όσον αφορά την εξαμηνία έκθεση για την ισότητα των φύλων. ή τέλο πάντων την αναδιατή έκθεση. Ε, να πω πάλι ότι συνοήθηκα με τους κοιοδησηγητές, να ευχαριστήσω πάλι την Μπλάνκα, την ε, Τζόρτζα αλλά και τη Γραμματεία. Με βοήθησαν για να συντάξω το κείμενο και θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική η δουλειά μας. Καλύψαμε πολλά θέματα και σημαντικά. αναλύσαμε τα στατιστικά δεδομένα, ό,τι είχε η έκθεση της ε, Κομισιόν. Είχαμε τις πληροφορίες από το Ίδρυμα ΕΓΕ. Είχαμε κάποιους δείκτες, κάποια στοιχεία. Είπαμε ότι υπάρχει εξέλιξη έστω και αργή. Σε άλλα μέτωπα βέβαια τα πράγματα ε, χαρακτηρίζονται από πισωγύρισμα. Και είπαμε ότι υπάρχουν ε, σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και γι' αυτό και είπαμε να ε, έχουμε μια νέα προσέγγιση, να δούμε τις επιδόσεις των κρατών μελών και πρέπει να γίνει σχετική συζήτηση ούτω ώστε να είναι επικοδομητικό το έργο μας και επίσης να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΓΕ λοιπόν 52,9 στα 100 είναι ο σχετικός δείκτης. Και σχέση με το 2005, δηλαδή, έχει ανέβει ο δείκτης κατά 1,5 μόνο, 1,5 μόνο μονάδα. Άρα, θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν ανισότητες σε πολλούς ε, τομείς. Επίσης, έχουμε και την ε, λιτότητα που δεν βοήθησε καθόλου, μάλλον χειροτέρεψαν τα πράγματα σε πολλούς τομείς και έχουμε το κενό, το χάσμα, το μισθολογικό στο 40%, το, τις συντάξεις επίσης είναι μεταξύ 11 και 36% των γυναικών που δεν έχουν καν πρόσβαση σε σύνταξη και οι νέες γυναίκες που δεν έχουν δουλειά είναι διπλάσιες από τους αντίστοιχους νέους νεαρούς άντρες. Πολύ ενισχυτικά όλα αυτά τα στοιχεία. Εάν τώρα δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, της ε, λιτότητας, τότε θα καταλήξουμε ότι οι γυναίκες χτυπήθηκαν περισσότερο από όλους από την κρίση. Και όσον αφορά την υγεία, γενικές υπηρεσίες ε, και λοιπά, αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν φυγεί κυρίως έδειξαν τα αρνητικά του τις γυναίκε. άρα αυτά θα πρέπει να μα προσκολουθούν επιγόντω. Ο Επομένω. είναι πάρα πολύ σημαντικό στην έκθεση να τα πούμε όλα αυτά και λέμε ότι η διάσταση του φίλου ξεχάστηκε όσον αφορά τις περισσότερες πολιτικές που ασκήθηκαν. Άρα, όσον αφορά τις πολιτικές συστάσεις τη ε, έκθεση να σα πω με δυο λόγια ότι χρειάζεται ε, ενώ για το 2020 να υπάρξει ο, ο άξονας, ο πυλώνας για τη διάσταση του φύλου. Επίσης να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια που το ήδη το κάνουμε στην Επιτροπή μας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα πρέπει επίσης να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια, δείκτες για την ισότητα, σύστημα εποπτείας, παρακολούθησης, ε, δημοκρατία, θεμελιώδη δικαιώματα, κράτος δικαίου και επίσης να ε, υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για τη διάσταση του φύλου. Α, και αυτό να λαμβάνεται υπόψη σαν προοικοδότηση σε κάθε καινούργια πολιτική. Επίσης στην έκθεση τονίζουμε το τι γίνεται όσον αφορά τη διάσταση του φύλου που είναι κάτι το οποίο γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό και αυτό το συζητούμε πάγια σε σχέση με την ακολουθητία στρατηγική και τονίζουμε ότι ανησυχούμε για το πόσο ε, σε κάποιες πολιτικές ε, δεν λαμβάνεται αρκετά υπόψη η του φίλου και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν θα με αλλά εν κατακλείδη να σας ε, πω το εξή. Μελετάμε τα νομοθετήματα που υπάρχουν. Είπαμε με το 2017 να υπάρχει νομοθετική δέσμη προβλάσης κομισιών. Είπαμε ότι έχει γίνει κύρωση της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, Επίση υπάρχει και η σχετική οδηγία που είναι πολύ σημαντική και άλλα κατεπήγοντα επίσης υπάρχουν ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα των ε, προσφύγων από πλευράς του τι γίνεται με τις ε, γυναίκες. Επίσης το δουλεμπόριο, η εμπορία ανθρώπων. γιατί εδώ ε, υπάρχει το θέμα των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων στην υγεία. Και τέλος, είχαμε χθε εδώ την Διευθύντρια της ΕΓΙ να την ευχαριστήσουμε ε, γιατί μας βοήθησαν πολύ από σε ΕΓΙ για την έκθεση. Είναι ένα ίδρυμα πολύ αξιόλογο. Θα πρέπει να το προστατεύσουμε, να το υποστηρίξουμε. Το κάνουμε αυτό στο κείμενό μας. Επίσης, άλλη μια σημαντική σύσταση. Να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό για τους διάφορους μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν. Από πλευράς Κομισιόν, από πλευράς ΕΓΕ, τι κάνουμε με τους δείκτες, τι κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλύτερο συντονισμός θα πρέπει να γίνει. Ευθυγράμμιση. Ε, έχουμε ενιαίο χρονοδιάγραμμα κατά κάποιο τρόπο. Εδώ θα βγω τελεία. Νομίζω ότι στο κείμενό μας καλύπτουμε πολλά ζητήματα και ευχαριστώ να αρχίσω τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρία Ζοβάρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά γιατί λέω δεν υπάρχει διερμηνία από τα τσέχικα, από τα τσέχικα μάλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή, τον συνάδελφο τον κ. Ουρτάσον, ε, για την έκθεση αυτή που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι πολύ καλά δομημένο. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σε εμπεριστατωμένα στοιχεία είναι σημαντικό να μην μπούμε σε μια ιδεολογική προσέγγιση και να είμαστε συγκεκριμένοι. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε συνένεση. Βεβαίως η κατάσταση των γυναικών σε σχέση με τις, ε, τις διαφορές τους μισθούς, τις συντάξεις, ε, δεν είναι η καλύτερη. Δεν είναι επαρκής η κατάσταση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά την θέση των γυναικών στις χώρες της Ένωσης για τα ζητήματα αυτά. Η έκθεση λέει κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Λέει ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών η σχετική πολιτική είναι όλο και λιγότερο σημαντική. Δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη στις πολιτικές των χωρών το θέμα, για το θέμα αυτό. Εγώ νομίζω ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δηλαδή έχετε επαρκή στοιχεία για να το πείτε αυτό, θα πρέπει να αναζητήσετε, να αναζητήσουμε, γιατί η, αλλαγή, η πολιτική για το θέμα των δύο φύλων ε, παραμερίζεται γιατί δεν ε, έχει επιτυχία. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε, να το σκεφτούμε το θέμα αυτό. Ίσως ορισμένε φορές να ε, καταφεύγουμε υπερβολικά στην ιδεολογία. να, δηλαδή να αναφέρεται ίσως όταν διοφύλουν σε όλες τις πολιτικές. Ίσως να μην είναι η σωστή προσέγγιση. Ίσως να πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στα σημεία που έχει πραγματικά σημασία. Πάντως σας ευχαριστώ που περιγράψατε την κατάσταση αυτή. Είναι σημαντική. Ε, είναι σημαντικό ότι το κάνετε, είναι σοβαρή η κατάσταση. Θα προετοιμάσω τροπολογίες πρέπει να βρεθεί συνένεση, θέλουμε να βρεθεί συνένεση, έτσι ώστε η έκθεση στην τελική της μορφή να συνεισφέρει πραγματικά στην αναζήτηση της βελτίωσης της κατάστασης για το θέμα της ε, απόκλησης ε, των, του επέδου συντάξεων. Ε, οι αναφορές τώρα στα δικαιώματα τα αναπαραγωγικά στην έκθεση νομίζω πως δεν είναι αναγκαίες. Θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίες. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να αναφέρουμε αυτά τα ζητήματα αυτά σε όλες τις εκθέσεις. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την προσέγγισή σας και αναμένω τη συζήτηση που θα γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο για το θέμα αυτό. Εάν όχι, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ήθελα απλώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ε, μια κοινή ε, διάγνωση της κατάστασης με βάση συγκεκριμένα περιστατωμένα στατιστικά στοιχεία και σε τακτική ε, σε τακτικό χρονικό διάστημα. Εμείς κάθε χρόνο το Μάρτιο, κοντά δηλαδή στην 8η Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας, ε, δημοσιεύουμε μια έκθεση και έχουμε τρεις στόχους με την έκθεση αυτή. Ε, θέλουμε να εξετάσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τις τάσεις ε, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, να έχουμε μια, μια κοινή διάγνωση. Θέλουμε να εξετάσουμε τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου υπάρχουν δράσεις ε, για την ισότητα των δύο φύλων, στον τομέα της έρευνας, ε, του αθλητισμού επίσης ε, και ο στόχος της έκθεσης είναι επίσης να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, να παρουσιάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη ή κάποια project που πραγματικά να έφεραν αποτέλεσμα διάφορα project, προγράμματα που προέρχονται από κάτω ε, και τα οποία έχουμε εμείς ε, χρηματοδοτήσει και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευση για όλους τους εμπλεκόμενους ε, στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ντεβουάν. Ο Έρνεστ για να κλείσει τη συζήτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ Ζωάο. Θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κυρία Γιώροβα. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και διμερώς. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους ε, υπάρχει μείωση του ειδικού βάρους ε, της ε, πολιτικής ισότητας ε, στις ευρύτερες, στον ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό των κρατών μελών της Ένωσης και να δούμε βέβαια τι μπορούμε να κάνουμε για να το αναστρέψουμε. Αυτό να το βελτιώσουμε. Είμαι έτοιμο να συζητήσω μαζί σα. Ε, είναι ένα σημαντικό θέμα. Τώρα βεβαίω το θέμα των αναπαραγωγικών ε, δικαιωμάτων ε, το έχουμε συζητήσει. Είναι σημαντικό θέμα για την ομάδα μου. Αυτό που έχουμε συμπεριλάβει στην ομάδα, στην έκθεση, ε, δεν λέμε τίποτα που να μην έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, έτσι. Ε, Εν πάση έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ και είμαι, στη διάθεσή σας να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να, μάλλον να, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους, συγγνώμη. Ε, μάλιστα. Έχουμε και τη σκιώδη εισηγήτρια ε, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Παρακαλώ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση μόλις έφτασα υπήρξε καθυστέρηση στο αεροδρόμιο και δεν φταίω εγώ γι' αυτό ήθελα όμως να βρεθώ εδώ σήμερα ήθελα να συνεισφέρω κι εγώ διότι είναι σημαντικό το θέμα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, βεβαίως, τα τελευταία χρόνια. Όμως, καμία, σε καμία από τις χώρες μας δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις. Βεβαίως, παγκοσμίως η Ευρώπη ε, συγκριτικά είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και βεβαίως υπάρχουν διαφορές και εντός της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη ακολουθούν διαφορετικές ε, πολιτικές, ε, έχουν διαφορετικές δομές. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το δούμε. Κάποιες χώρες έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από άλλες. Και εδώ υπάρχει απόκληση. 55% των πολιτών της Ένωσης θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση στον τομέα αυτών. Τα κράτη-μέλη όμως είναι υπεύθυνα για τους τρεις βασικούς τομείς όπου η ισότητα των δύο φύλων ε, έχει τη σημασία της το τομέα της εκπαίδευσης, ε, της φορολογικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας. Ε, είχαμε φτάσει σε συμφωνία για κάποια από τα ζητήματα αυτά επί τη αρχή πριν από μερικά χρόνια και γενικότερα με την έννοια της ε, συμπέριληψης των γυναικών στις πολιτικές αυτές. Ήταν κάτι το οποίο πριν από 20 χρόνια ήδη είχαμε πει ότι θα συμπεριληφθεί στις πολιτικές μας. Όμως ε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά με πολύ ψηλά επίπεδα φτώχειας ε, στις γυναίκες, ιδιαίτερα ε, στις μονογονεϊκές οικογένειες που συνήθως είναι η γυναίκα βεβαίως ε, η μητέρα και ε, βεβαίως το σύστημα του κράτους πρόνοιας ε, δεν δίνει επαρκή στοιχεία στις γυναίκες τα, τα τα δικαιώματα αναπαραγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βεβαίω, συνήθω αυτό ε, συνοδεύεται από υψηλή ανεργία. Και οπότε έτσι υπάρχει πραγματικά πρόβλημα ε, ευάλωτη θέση στην αγορά απασχόληση. Και πέραν όλων αυτών θα πρέπει να προσθέσουμε τα εξή. Είναι το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Και ακόμα και όταν ε, δεν υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα καταγραφής των τόσων προβλημάτων στα κράτη-μέλη. Έχουμε αυτή την κατάσταση και εμείς εκπροσωπώντας τους Ευρωπαίους θα πρέπει να βρούμε ε, μια απάντηση μια απάντηση ενιαία, μια διεύθυνση που να προσφεύγουν όλοι και αυτό να το βάλουμε στην έκθεση για την οποία ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του. Είναι πλήρης η έκθεση. Είναι προοδευτικό αυτό το κείμενο που καλύπτει όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα που σας είπα. Νομίζω ότι εξαντλητικά φύγει ένα προς ένα τα ζητήματα και τα προβλήματα. Βέβαια ε, έχουμε και τις εκθέσεις του 14 και του 15 αλλά θέλω να σταθώ ακριβώς στο θέμα της βίας κατά των γυναικών. Και επίσης να ασχοληθούμε και με την Ιντερνετική βία, αυτό που λέμε κυβερνομπούλινγκ. Αυτό σοβεί και στην Ιταλία, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας. Και πρόκειται για κάποια κορίτσια πολύ νέα που πέφτουν θύματα αυτής της ε, πρακτικής. πρόσφατα Είχαμε και μια περίπτωση που συζητήθηκε πολύ από τον κόσμο γιατί κατέληξε σε αυτοκτονία ε, ενός κορισιού σε συνέπεια αυτού του κύβερνο bullying. Άρα θα πρέπει αυτό το θέμα να το αναδείξουμε. Το πώς κορυφώνεται αυτό το μίσος και τις ε, γυναίκες σε κοινότητες, σε σχολεία. Ε, πρόκειται για κάποια στρεβλή, διαστραμμένη νοοτροπία. Οπότε και εδώ μπαίνει το θέμα της ισότητας των φίλων, γιατί πολύ συχνά λέμε ότι ε, αναμφίβολα πρόκειται για ένα δικαίωμα που παλεύουμε να αναγνωριστεί, κάτι το οποίο εδώ και δεκαετίες αφορά τους αγώνες μας. Το πώς, επομένως, το χάσμα των δύο φύλων πρόκειται να γεφυρωθεί. Να δούμε επίσης το πόσο αν αυτό το χάσμα, αυτή η διαφορά, θα ωφεληθεί η ανάπτυξη και η οικονομία και γι' αυτό άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα υπάρξει πιο δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων στο σπίτι, στον νοικοκυριό. Είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα, το έχουμε πει και στην Κομισιόν. Πρόκειται για δουλειά που δεν αμείβεται. Και επίσης όλες οι υποχρεώσεις των γονέων τελικά καταλήγουν να τις φέρουν στις πλάτες τους οι γυναίκες. Άρα θα πρέπει να δούμε τα θέματα το, της όντας των δύο φύλων που θα πρέπει να εμπνέουν όλες τις στρατηγικές. Αυτό θα πρέπει να προσέξει η Κομισιόν. Ε, κατακλείδη και πάλι να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Πάρα πολύ καλή ήταν η δουλειά του και πιστεύω ότι μαζί θα μπορέσουμε έτσι να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, προς την ισότητα που θέλουμε, που ελπίζουμε να συμβεί. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Έρνεστη. Θες να αστρολογήσεις, ορτάσουν. Ευχαριστώ την συνάδελφο για όσα είπε. Βεβαίω και συμφωνώ με όσα μα εξήγησε η κυρία Πιτσένο. Και αν μα είπε τι γίνεται με τα θέματα τη ε, απασχόληση, με τα θέματα της βία. Ναι, αυτά προσπαθώ να τα θίξω. Α, είναι και το θέμα του κυβερνομπούλινγκ και αυτό μπορούμε να το καλύψουμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού βίου και ιδιωτικού βίου και κλπ. Και πάλι να ευχαριστώ την κυρία Πιτσένα Πολύ παραγωγική συνεργασία μας στις συναντήσεις ε, των σκιωδών. Ωραία, ολοκληρώσαμε και αυτό το θέμα. Οπότε, σας ενημερώνω ότι για τις ε, τροπολογίες. Η προθεσμία είναι η 18η Οκτωβρίου. τότε να τις έχετε υποβάλει. Δεν θα πω στους που παρίστανται το εξή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε τα επόμενα δύο θέματα. Δεν θα συζητήσουμε γιατί λείπουν οι εισηγητέ. Άρα ας πάμε στο τελευταίο θέμα για την ε, πρωινή μας συνεδρίαση. Γιατί είναι εδώ η Μαρία Ρενά. Ας συζητήσουμε αυτό επομένως. Γιατί αυτή η περίπτωση βέβαια θα πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά στην ημεσαριάταξη. διάταξη. Αλλά βέβαια κάποιοι σκιώδες ε, είχαν υπόψη τους ότι αυτό το θέμα της Μαρία Ρενά θα πάει στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης και δεν είναι εδώ. Επομένως, ή θα πρέπει να κάνουμε ένα 15 λεπτό διάλειμμα και να περιμένουμε τους ε, συναδέλφους για τις άλλες ε, ε, εκθέσεις, ας πούμε την κυρία Λεγκρίπ, ή να συζητήσουμε το άλλο θέμα που έχει μείνει, όπως είχαμε αποφασίσει δηλαδή. Τι λέτε, αρενά. Δεν έχω πρόβλημα, λέει η κυρία Αρενά. Ας συζητήσουμε όπως είχαμε πει το τελευταίο. Αλλά βέβαια το θέμα είναι αν είναι εδώ οι σκιώδες συγκητές. Δεν έχω πρόβλημα εδώ.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 θα είμαι σύντομη και βεβαίω αναμένω και τις τροπολογίες για αυτούς τους Ευρωπαϊκού πυλώνες των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό νομίζω, ναι, με ακούτε ναι, είναι σημαντικό ε, να μπορέσουμε να συζητήσουμε στην Ευρώπη το θέμα αυτό και τη δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της απασχόλησης. Ε, εκεί έχουν συμπεριληφθεί αυτές οι προτεραιότητες που είναι προτεραιότητες που σχετίζονται με το φύλλο. Ε, θα αναφερθώ σε δύο προτεραιότητες που υπάρχουν ήδη σε αυτά που έχουν γίνει στον τομέα της, απασχό... της απασχόλησης και μας ε, αφορούν βεβαίως άμεσα. Είναι σημαντικό να έχουμε δείκτες ε, με βάση το φύλλο που να μας επιτρέπουν να εξετάζουμε την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών των κοινωνικών δεύτερον νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις για την ε, ισορροπία μεταξύ της εργασιακής ε, ζωής ε, και της προσωπικής ζωής, την επανεξέταση της οδηγίας ίσης μεταχείρισης στην αγορά εργασίας και αυτά αποτελεί βέβαια προτεραιότητα για μας και τέλος η προτεραιότητα που έχει να κάνει με τις κοινωνικές επενδύσεις όπως η ύπαρξη ε, μιας εγγύησης ε, για τα παιδιά μέσω του ΦΕΝΤΕΡ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, διότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική ζωή και προσωπική ζωή σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν υποδομέ, υποδομέ υποδοχή ε, για τα μικρά παιδιά, παραδείγματο χάρη, έτσι ώστε οι κοινωνικέ επενδύσει να μπορέσουν να τύχουν υποστήριξη από τα Διευθυντικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ακόμα και αν αυτή η έκθεση περιλαμβάνει αυτά, αυτές τις προτεραιότητες, ε, αυτά υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθεί αυτή η έκθεση όσο έχει αυτή τη στιγμή επί τεσσάρων σημαντικών σημείων. Το πρώτο αφορά το θέμα των πιο ευάλωτων ανθρώπων, η καταπολέμηση της φτώχειας και ιδιαίτερα των μονογονεϊκών γονεϊκών οικογενειών, το θέμα της ενίσχυσης της εγγύησης των παιδιών Child Guarantee σε σχέση με την φτώχεια και εδώ, δηλαδή να πούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εξαιρώνται κοινωνικά, πολιτιστικά. Μιλάμε συχνά για τις ε, υποδομές ε, υποδοχής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Ε, εδώ μπαίνουμε σε φαύλους κύκλους φτώχεια. Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, που δεν έχουν πρόσβαση ε, στην κοινωνία, που δεν έχουν πρόσβαση στον, ένα ζεστό γεύμα μια φορά τη μέρα, ε, αυτά τα παιδιά ε, ε, πέφτουν στη φτώχεια και πρέπει αυτό το θέμα να το έχουμε κατά νου. Ένα άλλο θέμα τώρα. Πρέπει να, είμαστε, να επιμένουμε περισσότερο στο θέμα της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασία. δεν είναι μόνο θέμα της γονικής άδειας, της άδειας μητρότητας, είναι το θέμα της ίδιας της πρόσβασης της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Εδώ πρέπει να δώσουμε έμφαση. Επίσης, ε, στα εκτιμώντας της πρότασης ε, ε, γίνεται αναφορά στο θέμα του, της απόκλησης στην τομέα των συντάξεων, αλλά δεν υπογραμμίζουμε αρκετά το θέμα αυτό. Για μένα είναι σημαντικό να το εξετάσουμε ως θεμελιώδες μέρος, ε, θεμελιώδες πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, δικαίωμα στη σύνταξη λοιπόν, συντάξεις όμως που να μην είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι και αυτό μια προτεραιότητα την οποία θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, εμείς στην Επιτροπή Γυναικών. Ε, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε. Από εκεί πέρα έγιναν κάποιες προτάσεις, ε, τροπολογίες που να αποβληθούν έως τις 13 Οκτωβρίου, η ψηφοφορία θα γίνει 8 και 9 Νοεμβρίου ε, και τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, απασχόλησης τον Δεκέμβριο. Είμαι ανοιχτή και αναμένω τις προτάσεις σας για βελτίωση της, ε, του κειμένου που έχουμε μπροστά μας. Ε, μάλιστα, ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Τώρα, επειδή λείπουν πολλοί από τους σκιώδεις εισηγητές, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να μιλήσει από το ΕΛΚ. Μάλλον όχι. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ ω κοιόδης εισηγητή για την έκθεση αυτή. Σε σχέση με το αρχικό κείμενο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε κάποια θέματα που ακούσαμε στην εισαγωγή, κάποιες ανησυχίες Στην Επιτροπή Απασχόλησης ήδη έχουμε επιφυλάξεις και τις έχουμε δηλώσει αφορά την εφαρμογή του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων γιατί θα πρέπει πρώτα να το έχουμε αναλύσει ναι μεν έχουμε κάνει μια ανάλυση αλλά θεωρούμε ότι θα είναι ουσιαστικά πιο πολύ διακοσμητικός ο ρόλος, δεν θα είναι ουσιαστικός. Και επίσης και τα ερωτήματα που συνδέονται και έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά ε, δικαιώματα, που θα πρέπει να απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα. Κάτι άλλο που μας απασχολεί είναι η προσπάθεια εναρμόνισης ειδικά σε συγκεκριμένες χώρες όπου όπου οι κοινωνικές ε, διατάξεις ε, για το εργασιακό δίκαιο κτλ. είναι πολύ παγιωμένες. Αυτό όσον αφορά την πρόταση για την ε, δημιουργία πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα αντιξαχθεί μεγάλη συζήτηση στην Επιτροπή Απασχόληση και θα συνεισφέρουμε και εμεί αυτή τη γνωμοδότηση φυσικά. Δεν γνωρίζω αν κάποιο από τους ε, πράσινου θα ήθελε να πάρει την, ε, το λόγο. Επομένως, θα οδηγηθούμε στα συμπεράσματα όταν έχετε να κάνετε κάποια άλλα σχόλια. Μέχρι 17 Οκτωβρίου έχετε περιθώριο να υποβάλλετε τροπολογίες για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε στα άλλα δύο θέματα της μερικής διάταξης καθώς η Κωνσταντς Λεγκρίτ είναι εδώ μαζί μας φαντάζομαι ότι είναι έτοιμη να παρουσιάσει την έκθεση για την ανάγκη μια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάργηση και την αποτροπή των συνταξιδοτικών ενισοτητών λόγω φύλου, λόγω στην Κωνσταντς. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à, à chacune et à chacun d'entre vous. Euh, d'avoir euh, peut-être. Euh, σας ευχαριστώ όλους και σας πρόεδρε. Ε, κάπως ανακατεύθηκαν τα θέματα στην μέση διάταξη, αλλά τέλος πάντων. Εδώ είμαστε και έτσι μπορούμε να κάνουμε την ανταλλαγή ε, απόψε. Να σας πω τι γίνεται με αυτή την ε, έκθεση που ανέλαβα μετά το καλοκαίρι, αλλά βέβαια και πριν τις διακοπές είχαμε κάνει μια ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο σας είχα στείλει και ήταν θετική η τοποθέτησή σας επ' αυτού ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις, συναντήσεις, οπότε και έχουν διαμορφωθεί για μένα κατευθυντηρίες γραμμές για αυτή τη δουλειά. Τώρα, σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές ανισότητες. πρώτη για 38% αυτό είναι το νούμερο. Δηλαδή 38 ευρώ στα 100. Για κάθε 100 είναι 38 ευρώ η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 2013 μετρήθηκε αυτό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 38% Ε, βέβαια αυτό είναι πολύ ανησυχητικό πως καταλήξαμε εκεί γιατί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση γιατί αυτό δεν είναι αρκετά γνωστό και για αυτό η πολιτική μας ομάδα πρότεινε στην Επιτροπή μας να αναλάβει το θέμα, να διαμορφωθεί μια συνένεση και να μπορέσουμε να δούμε πώς σε κάποια φάση θα ελκύσουμε την προσοχή του κόσμου στο πρόβλημα, σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό το ζήτημα αυτής της μεγάλης ανισότητας, που είναι κάτι το οποίο αφορά όλα τα κρατη Επομένως, ανισότητα στην σύνταξη μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία κάποιου. Βέβαια είναι και θέμα αμοιβή, γιατί οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο. Και βέβαια υπάρχουν και οι διακοπές στη σταδιοδρομία. Αυτό αφορά πιο συχνά τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Για λόγους οικογενειακούς γίνονται αυτές οι διακοπές βεβαίως και αφορά τη μητρότητα, βεβαίως και το θέμα αυτό οδηγεί επίσης και σε ε, εργασία part-time, οπότε όλα αυτά αποτελούν εξηγήσεις γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο της συνταξιωτικής ανισότητας. Επίσης, είναι και θέμα της μεθόδου υπολογισμού. Είναι θέμα συστήματος συνταξιοδοτικού. Πολλές φορές οδηγούμαστε σε μια παγίδα παινίας ε, όσον αφορά τη σύνταξη. Και αυτό το φαινόμενο φύγει περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Όπως είπαμε, αυτό είναι κάτι το δυσάστοτο, το ενισχυτικό. Έχουμε στο κείμενο αυτό, τα βασικά του εγγράφου εργασίας που πριν τις διακοπές σας είχα υποβάλει και προσπαθούμε να φωτίσουμε το θέμα γιατί είπαμε ότι έχουμε εδώ πολλές μεταβλητές του προβλήματος των ανισοτήτων αυτών ανδρών και γυναικών το θέμα είναι τόσο τερατώδες που και οι ειδικοί δεν μπορούν να το συλλάβουν ε, συνολικά. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα το κατανοήσουμε καλύτερα, πώς θα το περιχαρακώσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να έχουμε στοιχεία, δεδομένα, συγκρίσιμα. Και βέβαια να αφορούν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ελπίζουμε ότι διάφοροι φορείς ε, και τα ιδρύματα τα οποία ασχολούνται με τις ανισότητες ανδρών θα μπορέσουν με αυτά τα στοιχεία κάτι να βγάλουν. Και στη συνέχεια να έχουμε συστάτευση όλων των ειδικών και να δοθεί μια απάντηση αποτελεσματική ούτω ώστε να φωτιστεί το θέμα, ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και αυτό να ξεκινήσει από τις ίδιες τις γυναίκες να βρεθεί απαρχή των λύσεων των δυνατών ούτως ώστε να βγούμε από αυτό το έξοδο των ανισοτήτων. Τα τρεις άξονες δράσεις μπορούν να επισημανθούν. Να δούμε πώς θα αξιολογήσουμε ό,τι ήδη ε, γίνεται, πώς μπορούμε να έχουμε και επιπλέον δράσεις σε νέα μέτωπα πλευράς Ευρώπης. να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, να μειωθούν αυτές οι ανισότητες όσον αφορά επίσης ε, το σύστημα των εισφορών γιατί πολλές φορές ακριβώς το ίδιο το σύστημα οδηγεί σε ανισότητες άρα και εκεί να συρρυκνώσουμε τις διαφορές και ανισότητες και επίσης να μειώσουμε τις ανισότητες επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της ταχυδρομίας οπότε θα πρέπει να έχουμε και επανεξιολόγηση των στρατιωτικών συστημάτων. Αυτό που ονομάζουμε gender gap, χάσμα των δύο, μεταξύ των δύο φύλων. Τώρα, πάρα πολλές είναι οι δυσμενείς διακρίσεις σε όλα τα συνταξιωτικά συστήματα. Και είπαμε ότι υπάρχει ανισότητα στις εισφορές γιατί υπάρχει ανισότητα και στους μισθούς. Τα ξέρουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Και είπαμε ότι είμαστε στο 16% για αυτή την ανισότητα και αν θέλουμε να άρουμε ε, αυτές τις διαφορές στις συντάξεις θα πρέπει πρώτα-πρώτα να φροντίσουμε για ε, την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων στο μισθολογικό. Είπαμε επίσης για την ε, διαδρομή, την επαγγελματική, τη σταδιοδρομία, τα θέματα που θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν. Έχουμε ευαισθησία σε αυτά. Είπαμε, έχουμε την κυρία Γιούροβα, την ε, επίτροπο που έχει δεσμευτεί να ασχοληθεί με το ζήτημα, να παρουσιάσει μια δεσμή μέτρων, στοχευμένων, ε, αποτελεσματικών, ούτως ώστε να οδηγηθεί η κατάσταση σε όλα τα επαγγέλματα, σε περισσότερη ισότητα, σε περισσότερη συμφιλίωση οικογενειακό και επαγγελματικό βίο. Και θα πρέπει τα κρατημέλη να κάνουν και αυτά το καθήκον τους, ούτως ώστε ακόμα και ο ιδιωτικό τομέας να βοηθήσει στην άρση των ανισοτήτων. Τώρα, όσον αφορά τα συντεξιωτικά συστήματα, Ε, είναι εθνική αρμοδιότητα και όχι ενωσιακή. Είναι θέμα βέβαια ανταλλαγή ε, αριστερων πρακτικών. Ξέρουμε ποια είναι αυτή η μέθοδος άρα, τις επισημαίνουμε, τις καλύτερες πρακτικές και φροντίζουμε για την διάδοση αυτών. Και αυτό θα βοηθήσει να έρθουν ανισότητες. Επίσης, να προβληματιστούμε όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού. Αναθεώρηση συστημάτων, αξιολόγηση ταξιδιωτικών συστημάτων, στα κράτη-μέλη, πώς γίνονται επομένω οι υπολογισμοί, σε σχέση με τις λεπτομέρειες λειτουργίας του συστήματος, διαπιστώνουμε στο πού μειονεκτούν οι γυναίκες και έτσι να έχουν ε, κάποιες προτάσεις, κάποιες συστάσεις στα κράτη-μέλη για να κάνουν τις αλλαγές στο σύστημα έχοντας ευαισθητοποιηθεί στο πρόβλημα. Οπότε, κυρία Πρόεδρε, Καταληκτικά μπορούμε να πούμε ότι για το σχέδιο του κειμένου είπα να προσέξω, να στοχεύσουμε το ζήτημα που θέλουμε. Δηλαδή, να δούμε πώς θα υπάρξει περισσότερη ισότητα όσον αφορά τις συντάξεις. Ούτως ώστε και οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Είπα να αποφύγω τις ε, παγίδες και εγώ και οι συνάδελφοι που με βοηθήσανε γι' αυτό είπαμε από κοινού για το σχέδιο κειμένου να λάβουμε υπόψη το σύνολο των ε, στεξιωτικών συστημάτων. Ε, να μην δούμε μόνο τα συγκεκριμένα θέματα που μας απασχολούν ως Επιτροπή ζητημάτων της γυναίκας. Να δούμε τι αφορά τις γυναίκες. Γιατί ήδη η Επιτροπή μας έχει συζητήσει συναφή θέματα και δεν υποτιμώ το παρόν πρόβλημα. Αλλά έχουμε ήδη εξετάσει το θέμα της φτώχειας που χτυπάει τις γυναίκες, το πρόβλημα του συγκερασμού, του ιδιωτικού βίου σχέση με τον επαγγελματικό βίο, οπότε ε, να ληφθούν υπόψη όλα αυτά που έχει κάνει η Επιτροπή μας. Επομένως ούτε να υποβαθμίσουμε ούτε να υπερεκτιμήσουμε το θέμα της έκθεσης. Και επίση είπαμε να προσέξουμε σε αυτή την ε, έκθεση να μην είναι δέντρο, δηλαδή ο καθένας εκεί να πλασάρει οτιδήποτε αίτημα και διεκδίκηση μπορεί να τον απασχολεί στην Επιτροπή μας. Για τις τροπολογίες. Προθεσμία 20 δεκάτου. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων ξανά στην Επιτροπή μας στις 29 Νοεμβρίου. Και επομένως στόχος είναι να ψηφιστεί η έκθεση αρχές του επομένου έτους, ίσως 25 Ιανουαρίου. Οπότε, εν όψη αυτού του χρονοδιαγράμματος, ευχαρίστως να ανταλλάξουμε απόψεις και κυρίω με του κοιόδη ηγητέ από όλες τι πολιτικέ ομάδε και όλους τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να προβληματιστούμε σωστά και να καταλήξουμε σε κάποια κοινή θέση. Σα ευχαριστώ. Η πρόεδρο. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στου ε, υπόλοιπου ομιλητέ, η κυρία Νόιν πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Λαγκρίπα. Μας δώσετε μια πολύ καλή παρουσίαση. Θέλω να σημειώσω κάποια πολύ θετικά σημεία αλλά και κάποια πράγματα που λείπουν. Πολύ θετικό είναι ότι έχετε μια πλευρη προσέγγιση. Υπάρχει μια προσέγγιση σε πολλά επίπεδα Και κάτι άλλο που παρατηρούμε συνεχώς είναι ότι υπάρχουν ε, κάποιες συγκρίσεις που δεν γίνονται και θα πρέπει να βελτιωθούν αυτά στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τα δεδομένα. Πολύ σωστά σημειώσετε ότι το συνδεξιδοτικό χάσμα προκαλεί προβλήματα και ότι αυτό συνδέεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Τα δύο αυτά αφορούν πολλές φορές γυναίκες που έχουν προσφέρει πολλά στον εργασιακό τομέα. Υπάρχει, είναι ένα φιλελεγόμενο θέμα στο ε, Familien Partei ε, γιατί αυτό έχει επιπτώσει και στι γυναίκε, αλλά και στι συντάξει των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια συζητάμε για το γεγονός πώς η κρίση έχει επηρεάσει τι γυναίκες. Αλλά εδώ σημειώνεται ότι έχει αρνητική επιπτώση κρίση και στις συντάξεις. Είναι δύσκολο να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση για τις ε, γυναίκες και επίσης ξεκάθαρα αναφέρεται ότι ο αριθμός των παιδιών ότι οδηγεί στη φτώχεια κάτι παράδοξο γιατί τα παιδιά σε κάνουν πλούσιο, είναι ένας εμπλουτισμός για την κοινωνία αλλά όταν λέμε ότι τα πολλά παιδιά κάνουν φτωχές στις γυναίκες είναι κάτι πολύ δραματικό, πολύ τραγικό. Θα ήθελα να σημειώσω και κάποια άλλα σημεία που θα μπορούσαν να καταλάβουν περισσότερο χώρο. Κάνετε λόγο για τη φτώχεια α, στη μεγάλη για τους ηλικιμένους ότι τους αποκλεί κοινωνικά. Τους αποκλεί και από τα καταναλωτικά αγαθά αλλά και από τον πολιτισμό και την συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα. Αυτή η συμμετοχή έχει να κάνει και με τον πολιτικό τομέα και με τον ε, πολιτισμικό τομέα και είναι σημαντικό. Επίσης παρατήρησε ότι η κρίση είχε επιπτώσει στις ε, συντάξει των γυναικών, ίσως έπρεπε να αποσαφηνίσουμε ότι τα μέτρα λιτότητα που ε, εφαρμόστηκαν μετά την κρίση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά έχουν επιπτώσει στις συντάξει των γυναικών. Όχι μόνο η κρίση, αλλά τα μέτρα λιτότητα επηρέασαν αρνητικά. Αυτό πρέπει να αναφερθεί. Τα κριτήρια για τις μεταρρυθμίσεις ε, που λήφθησαν στα κράτη-μέλη ναι, είναι σωστά, αλλά πολλές φορές δεν ε, επηρεάσει τις γυναίκες. Όσον αφορά το όριο εξεδότησης ε, στη Γερμανία, ήταν σίγουρα μια πολύ καλή πρόταση αλλά με 44 χρόνια εισφορά ε, από την πλευρά των γυναικών, τι μπορούν να πάρουν πίσω ω ως σύνταξη με τόσα χρόνια, με τόσα λίγα χρόνια. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε ότι για τα παιδιά είναι υπεύθυνοι και οι άντρες. Δεν είναι υπόθεση μόνο των γυναικών ότι μόνο οι γυναίκες θα πάρουν την άδεια ανατροφής αλλά και οι άντρες έχουν ευθύνη πρέπει να καταρρύψουμε αυτά τα στερεότυπα ότι τα παιδιά αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες και τις δεσμεύουν για μια ζωή. Όμως υπάρχει πάντα και ένας βιολογικός πατέρας, υπάρχουν και πατέρες από κοινωνικής πλευράς που και αυτοί έχουν ευθύνη. Και οι ιδιώτες δεν είναι μόνο να εργάζονται, αλλά να φροντίσουν και για τα παιδιά. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια πιο δίκαιη ε, κατανομή στη συντάξη σε σχέση με αυτό. Σημαντικό σημείο ε, και αυτό. Άλλα τρία θέματα που θέλω να θίξω. Εξατομήκευση του στεξιδοτικού συστήματος είναι καλή πρόθεση που υπάρχει στην ε, Γερμανία, όμω ε, ε, δεν ξέρουμε πώ θα είναι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει και από ευρωπαϊκή πλευρά να δούμε ποια θα είναι η βασική σύνταξη. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πολύ σημαντικά τα σημεία που αναφέρατε στην έκθεση θα μπορούσαν να επεκταθούν λιγάκι, ε, να προτείνουμε κάποιες τροπολογίες για να έχουμε ένα σωστό, ε, μια σωστή πρόταση. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, το, το, το που θα έχουμε το τελικό, αλλά να έχουμε δίκαιη συντάξη της γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ. Όταν συζητούμε το ζήτημα αυτό, επειδή τα θέματα αυτά είναι οριζόντια, η συζήτηση της έκθεσης αυτής έπρεπε να εξεταστεί από κοινού με προηγούμενες εκθέσεις αυτή για την φτώχεια, για την ε, ε, ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής ζωής και προσωπικής ζωής. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν αναπόφευκτο. Το θέμα των συντάξεων σημαίνει ότι μιλάμε βεβαίως για τους ανθρώπους, τους συνταξιούχους σήμερα, αλλά και τους αυριανούς συνταξιούχους. Τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα. Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να αναφερθούμε στην ευρωπαϊκή πολιτική, ε, στις πολιτικές λιτότητας. Υπάρχει βεβαίως η ευθύνη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και τη κοινωνική λειτουργία που πρέπει να έχει ένα κράτος, τον κοινωνικό ρόλο. Όλα αυτά πρέπει να αποτυπωθούν στην έκθεση Τώρα υπάρχουν μια σειρά από κρίσιμες πτυχές που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές της μισθολογική μεταξύ και γυναικών. Σε ό,τι αφορά την αύξηση παραδείγματος χάρη του ελάχιστου μισθού, την αντιμετώπιση ε, της, επισφάλ, της επισφάλειας που αφορά κυρίως τις γυναίκες. Οι γυναίκες εδώ τιμωρούνται διπλά. Διότι η επισφαλής εργασία αφορά σε μεγάλο ποσοστό τις γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις συλλογικέ συμβάσεις, ε, ε, τις συνθήκες εργασίας. Πρέπει να προσπιστούμε ε, μια αρχή που υπάρχει εδώ και 100 χρόνια. 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ψυχαγωγία. Είναι ένα βασικό στοιχείο για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τι κοινωνικέ ανισότητε, αλλά και τι ανισότητε μεταξύ των δύο φύλων. Και από εκεί πέρα υπάρχουν ακόμα μια σειρά από σημαντικά θέματα. Η εγγύηση τη ελεύθερη της ελεύθερης, της, ελεύθερης πρόσβαση στην παιδεία, στην η υγεία, στις δημόσιες υπηρεσίες γενικότερα, η ανάγκη ε, να, παρέχουμε, να παρέχουμε συστήματα που να υπερασπίζονται, να προστατεύουν τις οικογένειες, να τις στηρίζουν στην ε, φροντίδα των παιδιών τους, ε, στη φύλαξή τους. Η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσει ένα κράτος επίσης ε, ε, για την αξιολόγηση των συντάξεων αυτή η αξιολόγηση πρέπει να συνδέεται με την ενίσχυση των κοινωνικών συστημάτων που έχουν δεχθεί μεγάλη επίθεση τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από χώρες, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία. Είχαμε μια μείωση της χρηματοδότησης που υποτίθεται ότι εγγυάται την ε, σταθερότητα του συστήματος Αυτό συνδέεται βεβαίω και με τα υψηλά ποσοστά ανεργία που υπάρχουν στι χώρε τη Ένωση. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ε, ένα μια καθολική δημόσια υπηρεσία που να τα αποκρίνεται στις ανάγκες ε, των πολιτών. Αυτές είναι μόνο κάποιε από τι ανησυχίε που έχουμε. Αυτή θα είναι η συνεισφορά μας και αναμένουμε προφανώς ότι θα υπάρξουν και ιδεολογικέ διαφορές μια σειρά από σημεία αλλά γι' αυτό τα συζητάμε. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και με τους κοιόδους εισηγητές. Ε, μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος Βουρτάσουν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια, την κυρία Λεγκρή, για την παρουσίαση. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια απόκληση 40% στις συντάξεις είναι ένας ε, από τους βασικούς παράγοντες ανισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την έκθεση του 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρει ότι αυτή, αυτό το χάσμα έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν έως και 36% των γυναικών που δεν έχουν καμία σύνταξη. Επίσης υπάρχει το θέμα των ηλικιωμένων γυναικών, εξαιρετικά σημαντικό αυτό, διότι στην ομάδα των γυναικών άνω των 65 ετών έχουμε 7% περισσότερο φτώχεια από ό,τι τις νεότερες, νεότερες γυναίκες ε, και αυτό βεβαίως συνδέεται σε μεγάλο βαθμό ε, και με τα μειονεκτήματα ε, που υπάρχουν σε συγκεκριμένε επαγγελματικέ αδειοδρομίε. Ε, κάτι που το οποίο θα θέλει να, θέλει να, επιμείνουμε η ομάδα μα τουλάχιστον. Ε, το, οι μεταρρυθμίσει των συνταξιδοτικών συστημάτων τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τι γυναίκε. Διότι μεταξύ άλλων, πολλέ από τι μεταρρυθμίσει αυτέ ουσιαστικά ε, τιμώρησαν την μερική απασχόληση, που συνήθω είναι απασχόληση γυναικών. Ε, γυναίκε δηλαδή που έχουν. Ε, ε συσσωρεύσει διάφορες ώρες ε, εργασίας ε, μερικής απασχόλησης όταν ε, με το νέο σύστημα τιμωρούνται εν περιπτώσει στη σύνταξή τους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε κυρίως τον πρώτο πυλώνα των συντάξεων, το δημόσιο συνταξιδοτικό σύστημα δηλαδή, που είναι αυτό που ουσιαστικά είναι πυλώνας βασικός του συστήματος πρόνοιας της Ευρωπαϊκής Ένωση, ε, του συστήματο ε, του κράτους πρόνοιας ε, και από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει επίση να ενισχύσουμε την άποψη ότι τα συνταξιωτικά συστήματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το, την αναπαραγωγική διαδικασία είναι κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη να υπάρχουν συνταξιωτικά συστήματα που να λαμβάνουν υπόψη τις επαγγελματικές διαδρομίες, τους τομείς εκείνους, τους κλάδους εκείνους όπου ε, εργάζονται κυρίως γυναίκες. Επίσης ε, η σημασία της εξατομίκευσης της ε, φορολόγησης σε κάποιες χώρες δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Πιμέντα να υπάρχει μια ελάχιστη σύνταξη αξιοπρέπειας ε, το θέμα επίσης της φορητότητας των συντάξεων ε, είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να μας να καλύψουμε. Αυτά είχα να αναφέρω από εκεί πέρα. Ελπίζω να έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε με την κυρία Λεγκρίφ και με τους υπόλοιπους σκιώδεις ε, συγγητές. Η κυρία Αρενά έχει το λόγο τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία, την κυρία Λεγκρίφ και τα διάφορα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης ε, για το θέμα των ατομικών συντάξεων. Μια διαδικασία που θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί μάλλον στις 31 Οκτωβρίου και με ανησυχεί κάπως αυτή η δημόσια διαβούλευση. Είπατε προηγουμένως προσοχή, ε, οι συντάξει δεν είναι θέμα αρμοδιότητας ε, της Ένωσης, όμως η Κομισιόν δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα να ξεκινήσει με διαβούλευση για μια αρμοδιότητα την οποία δεν έχει έτσι για ένα θέμα αρμοδιότητας ε, που δεν είναι αρμοδιότητά τη. Εφόσον η Κομισιόν λοιπόν επιτρέψει τον εαυτό τη να κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχουμε και το θάρρο να πούμε τι δυνατότητε έχουμε ε, να εργαστούμε στο, δια... στο ζήτημα των συντάξεων. Και νομίζω ότι έχουμε ένα εργαλείο όλου ιδιαίτερω το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των Εθνικών Σχεδίων Μεταρρύθμιση, έω τώρα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των Εθνικών Σχεδίων Μεταρρυθμίσεων, ε, βλέπουμε συστάσει που έχουν να κάνουν με το, ε, με το να πιεστούν τα κράτη-μέλη να κάνουν λιγότερα για τις συντάξεις. Εμεί θέλουμε στα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να υποχρεώνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα πράγματα για τι συντάξει, για τα εξωτερικά συστήματα, στον υποχρεωτικό πυλώνα και να κάνουν και περισσότερα πράγματα για τι γυναίκε. Και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να καταγγείλουμε το γεγονό ότι υπάρχει 36% απόκληση και ότι τα κράτη-μέλη ε, υποχρεούνται από τις τάσεις αυτές να καλύψουν το κενό αυτό, το χάσμα αυτό. Έχουμε εργαλεία ευρωπαϊκά που χρησιμοποιούνται κατά τη γνώμη μου με λάθος τρόπο προς τη λάθος κατεύθυνση και ως Επιτροπή Γυναικών εμείς πρέπει να, χρησιμοποιήσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση με συστάσεις σημαντικές. Αντί λοιπόν να λέμε ε, εντάξει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορούν να πληρώσουν μέσω συλλογικών συμβάσεων ε, διότι αναφερθήκατε στις εισφορές, έτσι, ε, αντί να πούμε μέσω συλλογικών συμβάσεων δεν τα καταφέρνουμε, ε, θα κάνουμε λοιπόν ατομικές ε, θυσίες με συστήματα συλλογικά κεφαλαιοποίησης ιδιωτικά, ατομικά. Και πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε αυτές τις ανισότητες. Εάν υπάρχουν ανισότητες στο δημόσιο σεξουαλικό καθεστώς, δηλαδή το ανταποδοτικό, πιστεύουμε, πιστεύω ότι αυτές οι ανισότητες είναι ακόμα μεγαλύτερες σε ένα σύστημα κεφαλαιοποίησης. Διότι το σύστημα κεφαλαιοποίησης ουσιαστικά ζητεί, απαιτεί να υπάρχουν επαρκή, ε, επαρκές εισόδημα για να μπορέσει κάποιος να τα αποταμιεύσει. Κάποια γυναίκα που δουλεύει με μερική απασχόληση και δεν μπορεί να αποταμιεύσει, δεν θα πάει προς, μια, προς ένα σύστημα ε, εξωτερικό μέσο κεφαλαίο Διότι όταν κάποιο στο τέλο του μήνα ε, πληρώνει πια με επιστοτική κάρτα τα ψώνια του, δεν μπορεί να, να πληρώσει ένα σύστημα κεφαλαιοποίηση. Οι ευάλωτε λοιπόν γυναίκε, λόγω των συμβάσεων εργασία του, δεν μπορούν να πάνε προ ένα τέτοιο σύστημα. Αυτή είναι η πρώτη διάκριση σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση. Το δεύτερο, η επαγγελματική κλάδη. Διότι υπάρχουν επαγγελματικοί κλάδοι που καλύπτουν μέσω λογικών συμβάσεων στήματα κεφαλαιοποίηση. Είναι συνήθω η πιο πλούσιοι πραγματική πραγματική κλάδη, ο τομέα τη χημία. Βεβαίω και καλύπτει συστήματα σε εξωτικά μέσω κεφαλαιοποίηση, διότι είναι πλούσιος κλάδο. Υπάρχουν όμω πολλέ γυναίκε που δουλεύουν στον τομέα τη χημία. Όχι. Δυστυχώ όχι. Αυτοί λοιπόν που πληρώνουν καλύτερα είναι οι πιο πλούσιοι. Το σύστημα κεφαλαιοποίηση λοιπόν το σύστημα κεφαλαιοποίηση τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαβούλευση αυτή. Να ενισχύσουμε τι ανισότητε. Ενισχύουμε τι ανισότητε και ενισχύουμε τι ανισότητε μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, και θα ήθελα αυτό να αναφέρεται στην έκθεση για να μπορούμε να πούμε σαφώ ότι η βασική μα, η πρώτη μα ανησυχία, είναι ο καθεστώ του πρώτου πυλώνα. Εάν ενισχύσουμε ένα σύστημα δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει αποχρεωτικά να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των γυναικών σε σχέση με τι διακρίσει τι οποίε βιώνουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Αρενά και τώρα η κυρία Κολόσκα έχει λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με χαροποιεί το γεγονό ότι έχουμε αυτή την ε, έκθεση για το στεξιδοτικό χάσμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένου του χάσματος, του μεγέθους του χάσματος. Και ότι το χάσμα αυτό οφείλεται στην ε, συσσόρευση όλων των ανισοτήτων που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Έχουμε λοιπόν το εργασιακό χάσμα και το γεγονός ότι οι εργαζόμενες γυναίκες, ειδικά στα δυτικά κράτη-μέλη, εργάζονται ε, με μερική απασχόληση και επιπλέον οι γυναίκες πολύ, ε, πολύ συχνά εργάζονται σε χαμηλού εισοδήματος επαγγέλματα, όπου υπάρχει αυτό το όριο, το πλαφόν, έχουμε το, την ανισότητα στους μισθούς, τις ανισότητες στους μισθούς και επίσης Κατά 40% ε, χαμηλότερη έχουν οι γυναίκε σε σχέση με του άντρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, επομένως, Επομένω, πρέπει να επαναλάβουμε και να τονίσουμε ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ε, τεράστιο πρόβλημα, θα πρέπει να εξετάσουμε τι αιτίε αυτού του τεράστιου εξωτερικού χάσματο. Είναι το τελικό αποτέλεσμα τη επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών Άρα αν η σύνταξη είναι χαμηλή, αυτό οφείλεται στο... στην επαγγελματική του ζωή. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις όχι μόνο στο συνταξιδοτικό σύστημα, θα μπορούσε να παρέχει κάποιο αποζημίωση στο συνταξιδοτικό σύστημα, όπω στην Πολωνία που έχουμε εξοδοτικές εισφορές που ε, πληρώνονται από τις ε, γυναίκες στο εξωτερικό τους ε, πλάνο κατά τη διάρκεια της ε, άδειας μητρότητας, αλλά πρέπει παράλληλα να δούμε και τις αιτίε του χάσματος αυτού που οφείλονται στην αγορά εργασίας. Γιατί το αποτέλεσμα οφείλεται στον τρόπο που κινούνται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και για πολλά χρόνια, όπως είναι γνωστό, οι γυναίκες είχαν διαφορετική θέση ε, σε σχέση με αυτές που εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας. Ε, αυτό το χάσμα θα διευρυνθεί, είχαμε 40%, αυτό θα αυξηθεί και θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να να δούμε τη συγκεκριμένη θέση των νεαρών γυναικών στην αγορά εργασίας οι οποίες διατρέχουν τον κίνδυνο να έχουν μπροστά τους ένα ακόμα μεγαλύτερο συντεξιδοτικό χάσμα σε σχέση με τις μεγαλύτερες γυναίκες. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το συντεξιδοτικό χάσμα είναι απόρρια της θέσης στην αγορά εργασίας των γυναικών Και γι' αυτό, για να το αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στην αγορά εργασία. Σα ευχαριστούμε. Κυρία Λεγκρίπ, ακούσατε του συναδέλφου. Η κυρία Λεγκρίπ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Ναι, είναι πολύ θετικό το ήταν η ποιοτική σημερινή συζήτηση. Ακούσαμε διάφορες ε, απόψεις, όλοι συνεισέφεραν, όλοι δώσανε κάποιες ε, ιδέες για το τι να κάνουμε. Όχι καθόλου δεν απογοητεύτηκα, πρόκειται για ένα θέμα ε, μας απασχολεί και θα θέλουμε να το σκεφτούμε, να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε αξιόλογη έκθεση της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι θεωρήσαμε ότι όλοι θα εργαστούν, όλοι θα ενδιαφερθούν για το ζήτημα αυτό. Όλες οι πολιτικές ομάδες. Ε, ακριβώς γι' αυτό και ήταν τόσο αποδοσούν καρπούς. και ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Ελπίζω όλα αυτά να αποδώσουν ε, καρπούς. Και θέλω να σας επαναλάβω το εξής. Δεν είναι θέμα απουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη διαμόρφωση των συνταξιδοτικών συστημάτων, αλλά πρόκειται για θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Αλλά βέβαια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και συγκεκριμένα η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να σέβεται αυτή την κατανομή των ρόλων και αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επικουρικότητα. Όμως, για συγκεκριμένα προβλήματα θα πρέπει να βοηθάμε να πέφτει το φως. Ε, ακριβώς εδώ πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ή είπαμε πάλι ότι δεν θέλουμε να έχουμε μια έκθεση ε, που να έχει λίγο απ' όλα. Να μην είναι σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα ε, στολίδια, με οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να καλύψει από τον τίτλο αυτόν να είναι στοχευμένη η έκθεση, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα που θέλουμε. Βεβαίω και ξέρω ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τον οριζόντιο χαρακτήρα των θεμάτων για όλους αυτούς τις ε, μεταβλητές που οδηγούν στο μισθολογικό χάσμα, στην μισθολογική ανισότητα. Αλλά λάβει υπόψη ότι είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Και έτσι θα είναι το κείμενο συλλογικού χαρακτήρα. Στοχευμένο. Και για το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Αυτά προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε και σας κύριε Αλεγκρίπ και όλους όσοι μίλησαν. Όπως είπε η συγκήτρια, 20 Οκτωβρίου στις 5 η ώρα λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα το πρωί. για τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η κυρία Γκαμπριέλ είναι η συγγύτρια και έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω αυτό το ζήτημα για τις γυναίκες στα κράτη ανατολικής εταιρικής σχέσης. Εκ των προτέρων, ευχαριστώ τους και οδησυχητές για τη συνεργασία. Η σταθερότητα στη πνιάζουσες χώρες είναι αυτό το οποίο θέλουμε για να υπάρχει ειρήνη και ευημερία και οι γυναίκες σχετικά με αυτό έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ε, αυτές οι χώρε να ενεργούν σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο, να σέβονται τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών, αλλά βέβαια για το ζήτημα τη ισότητα ανδρών και γυναικών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής τη εταιρική σχέση. Θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο. Η ισότητα ανδρών και γυναικών επίση τονίστηκε στο ότι είναι και θέμα συνεργασίας. Είναι πολλά υποσχόμενο στην ε, Ρήγα, στην εκεί συνάντηση, δηλαδή κορυφή το 2015. Και είπαμε ότι οι γυναίκες ε, ε, πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στον κοινωνικό οικονομικό βίο και επίσης να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό που λαμβάνει χωρί χώρες όπως αυτές. Η Αρμενία, Ζερμπατζάν, Λευκορωσία και Γεωργία. Αλλά η Μολδαβία και η Ουκρανία είναι χώρες που διαφέρουν πάρα πολύ μία από την άλλη. Και βέβαια ε, υπάρχει διαφορετική σχέση με την κάθε μία από αυτές τις χώρες. Ακριβώς γι' αυτό και έχουμε την αρχή της διαφοροποίησης όσον αφορά την ε, πολιτική γειτονία. Και επίσης ισχύει το naming and shaming, του να κατονομάζεται όποιος δεν κάνει αυτό για το οποίο έχει δεσμευτεί. Οπότε, ε, είδαμε ποιες είναι οι δυσκολίες στην αρχή, είπαμε να δούμε ε, ποιες είναι οι πρακτικές, ποια είναι τα προγράμματα τα οποία πρέπει να αποδώσουν οι καρπούς και είπαμε ότι ο, το να κατονομάζεται ο φταίχτης θα πρέπει να ισχύει και για τα θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. Οπότε, με λίγα λόγια να σας πω ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Πρώτα-πρώτα έχουμε μια σύντομη εισαγωγή και εδώ λέμε ότι αυτές οι χώρες ήδη έχουν στρατευθεί να βοηθήσουν ε, για να αρθούν οι ανισότητες και αυτό κατοχύνει και στο Σύνταγμα και στην ε, κοινή νομοθεσία υπάρχουν και εθνικά προγράμματα αλλά κυρίω ε, αυτά γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Μετά έχουμε έξι διαφορετικά κεφάλαια στην έκθεση. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και εδώ τονίζουμε το ότι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στον πουργό Γίγνεσθε οι γυναίκες αυτές τις χώρες, να συμμετέχουν στις αλλαγές, επίσης και στον οικονομικό βίο θα πρέπει να αρθούν οι μισθολογικές ανισότητες, ε, οι ανισότητες στην αγορά εργασίας, όλα αυτά αποτελούν συστάσεις, επίσης η βία κατά των γυναικών, ε, η οικιακή βία, Βεβαίω, βασικά θύματα είναι οι γυναίκε. Να οι δύο βασικοί άξονε. Επίση, ο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκε όσον αφορά την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Σε αυτό το τμήμα τη έκθεση τονίζουμε ότι σε πολλέ ζώνε εμπόλεμε ε, συγκρούσεων τέλο πάντων ε, βοηθούν οι γυναίκε. Τα είπαμε αυτά στην ακρόασή μα. Επίση, ε, άλλο θέμα σημαντικό είναι οι αξιόλογες πρακτικές πρώτα τα προγράμματα, τα έργα που χρηματοδοτούνται, συγχρηματοδοτούνται από κράτη-μέλη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι είπαμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε την θετική δυναμική για όλες αυτές τις ε, χώρες. Επίσης, η βοήθεια το, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίασης, στήριξη, βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στα πλαίσια αυτής μας της πολιτικής, αλλά και στα πλαίσια της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ισότητας των Φύλων. Περιμένω τις τροπολογίες και θα προσθέσουμε και άλλα θέματα όπως ας πούμε το θέμα γυναίκες και εκλογές, το Euronest, την προσθέμενη αξία του φόρουμ των γυναικών, το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και έχουμε και άλλα παραδείγματα από αξιόλογες πρακτικές συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα δικαιώματα και η ισότητα θα πρέπει να τελειώσουν αντικείμενο ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ένωση και αυτών των κρατών. Τα περισσότερα αυτά τα προβλήματα είναι κοινά. Τα έχουν και εκείνοι, τα έχουμε και εμεί. Οπότε αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να βοηθήσω για τα δικαιώματα και για την ε, ισότητα. Να είναι θέματα ψηλότερης, μεγαλύτερη προτεραιότητα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Και θα λάβω υπόψη ό,τι προτάσεις μου κάνουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κυρία Μπορζάν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφό μου την κυρία Γκάμπριελ για την εξαιρετική έκθεση. Υπάρχουν πολλές πτυχές που θα ήθελα να τονίσω εκ μέρους της ε, ομάδας των σοσιαλιστών. Πρώτα απ' όλα ε, είναι τροπολογίες, προτάσεις που έχουν να κάνουν ε, με το διαχωρισμό ιδιωτική και ε, δημόσια ζωής και τα επαγγέλματα. Πολλέ φορέ οι γυναίκε δεν έχουν την εκπαίδευση για οικογενειακούς λόγους όπως δηλώθηκε από την κυρία Γκάμπριελ στην έκθεση και επίσης παραμελούν τη δική τους καριέρα. Ενισχύουμε τις υποδομές στην ε, φροντίδα των ε, παιδιών, στο να υπάρχουν ε, παιδικοί σταθμοί, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να αφοσιωθούν στην εργασία τους, αλλά και για τους ηλικιωμένους, γιατί πολύ συχνά ηλικιωμένοι φροντίζονται πάλι από τις γυναίκες. Θα αναφερθώ σε διάφορα προγράμματα για την ενίσχυση της οικονομικής θέσης των γυναικών και τα συνδικάτα παράλληλα, όπως είναι πολύ σημαντική και οι μηχανισμοί μικροπίστωση όσον αφορά την ε, ελευθερία διακίνηση προσώπων, η καταπολέμηση της βίας στο πλαίσιο της οικογένειας, το ποσοστό αποδοχής της ενδοοικογενικής βίας είναι σοκαριστικό, γιατί δείχνει ότι θα πρέπει οι γυναίκες να το ανέχονται για να κρατήσουν την οικογένεια ενωμένη. Οι γυναίκες θα πρέπει να καταγγέλουν όλες τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και χρειάζονται ένα σύστημα υποστήριξη από ειδικού, από συμβούλους, από την αστυνομία και από ιατρικό προσωπικό. Πολύ σημαντική είναι η πρόσβαση σε αντισυλληπτικά σε περίπτωση ανηλίκων που παντρεύονται. Μα σοκάρει επίση η είδηση ε, για επίθεση ενάντια σε άτομα LGBT e στη δουλειά. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής είναι ότι υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και οι γυναίκες πρέπει να εμπλέκονται γιατί πολύ συχνά είναι θύματα αυτών των συμπλοκών, των σειράξεων. Αυτό αφορά και στα παιδιά βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο του σε ειρηνευτικέ ε, ε, αποστολέ. Επίση, έχουμε και τι γυναίκε που ετούνται άσυλο. Πολλοί θα μα βοηθήσουν να έχουμε μια ολοκληρωμένη έκθεση η οποία θα προωθεί θετικέ αλλαγέ ε, στι χώρε τη Ανατολική και των εταιρικής σχέσης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ποιοτική έκθεση. Προέρχομαι από χώρα που είναι κοντά στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Άκουσα αυτό που για την ανάγκη οθέτηση μια θετική προσέγγισης. Η έκθεση περιέχει σωστές παρατηρήσεις και αυτό που με ικανοποιεί είναι αυτό που υπόθηκε τη συμμετοχή ε, των γυναικών σε εμπνευστικέ αποστολέ. Κάτι που θα πρέπει να προωθηθεί. Οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι γείτονε θα πρέπει να διδραματίσουν ε, ένα πιο σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να εντατικοποιήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής ε, Σχέσης. να έχουμε ανταλλαγή εμπειριών ε, ώστε να αποκτήσουν ε, και αυτές οι χώρες την απαραίτητη εμπειρία και να δώσουμε προσοχή επίσης σε πρακτικά θέματα όπως είναι η προσβασιμότητα σε παιδικούς σταθμούς, σε χώρους για άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους και άλλες ε, ομάδες του πληθυσμού. Είναι ένα θέμα το οποίο θα δείξω και στην πρώτη τροπολογία. Ευχαριστώ κυρία Κολόσκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ ε, την εισηγήτρια για την εξαιρετική αυτή έκθεση. το βασικό εδώ είναι η εισαγωγή του mainstreaming σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να πείσουμε τους υπεύθυνους, τους κυβερνητικούς θύνοντες των χωρών αυτών, ότι το θέμα αυτό είναι όντως σημαντικό. Στις συζητήσεις με τη Δύση και στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις χώρες αυτές. Διότι αυτές οι αλλαγές στις χώρες αυτές, αυτές οι μεγάλες αλλαγές έχουν τις ήρωές τους ε, και μεταξύ των αυτών υπάρχουν και οι γυναίκες. Είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα της ίσης μεταχείρισης δεν πρέπει να μείνουν στην ανωνυμία ε, οι γυναίκες αυτές, αυτές να παραμείνουν ορατές επίσης ο ρόλος των γυναικών στην επίλυση διαφορών, στην επίλυση σειράξεων, όχι μόνο εξωτερικών σειράξεων με γείτονες, αλλά και οι εργαζόμενες ε, στην αστυνομία παραδείγματο χάρη και βεβαίω, ε, όταν αυτές οι υπηρεσίες ανοίγουν στι γυναίκες φαίνεται αμέσως η διαφορά και πρέπει να πω ότι στην Πολωνία το 2013 ε, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα ε, γυναικών που εργάζονται σε τέτοιου είδου υπηρεσίες με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων γυναικών που ξεκίνησαν κάποιες άτυπες ε, επαφές τελικά επισημοποίησαν ε, αυτή τη διαδικασία δημιούργησαν μια ομάδα η οποία συνδέεται απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και που εξετάζει τα προβλήματα που προκύπτουν σε διάφορες υπηρεσίες αυτές για τις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αστυνομία, στην, ε, στο να ενταχθούν παραδείγματος χάρη στην στις αστυνομικές υπηρεσίες, ε, υπάρχει μεγάλη πρόοδο, κάτι που δεν ισχύει ακόμα όμω στον τομέα του στρατού, παραδείγματο χάρη, ή τον τομέα τη πυροσβεστική. Χάρη ε, ε όμω ε, σε αυτή την πρωτοβουλία στην αστυνομία έχουμε ένα άνοιγμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια δικτύωση μεταξύ των γυναικών και νομίζω ότι το Euronest μπορεί να παίξει ένα ρόλο εδώ πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτό, πρέπει ε, να επεκταθεί. Να έχουμε δηλαδή εδώ άλλη μία ε, πρωτοβουλία που θα ενισχύσει τον ρόλο των γυναικών και τον ρόλο μπορεί να παίξουν στην ανάπτυξη των χωρών τους. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν η κυρία Γκάμπριελ θέλει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όχι, ήθελα απλώς ε, να σας ευχαριστήσω. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα σχόλια, τις προτάσεις, τις ιδέες. Θέλω να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω όλους, διότι χάρη στις δικές σας παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κείμενο αυτό, να εμπλουτίσουμε και να προωθήσουμε ε, τις απόψεις μας. 17 Οκτωβρίου ημερομηνία προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ολοκληρώνουμε σήμερα το πρωί. Ε, θα τα ξαναπούμε το απόγευμα στις 3.